Good afternoon, colleagues. A warm welcome. Καλησπέρα σας. Ε, να σας καλωσορίσω θερμά όλους και να καλωσορίσω θερμά και τον κύριο Τομάστε Τεμεζιέρ, Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και τον κύριο Ματάες Φέκλη, Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, ε, για ανταλλαγή απόψεων εδώ με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σχετικά με το διάλογο για την ασφάλεια. Όπως γνωρίζετε, έγινε ο πρώτος διάλογος μου για την ασφάλεια πριν από τέσσερις ημέρες με τον Επίτροπο Κίνγκ και επειδή επικεντρωνόμαστε τώρα σε αυτά τα θέματα, θα συζητήσουμε με τον δύο υπουργού από τη Γερμανία και τη Γαλλία. Όπω γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έχουμε τακτικέ επαφέ με την Προεδρία. Κάθε εβδομάδα είμαστε σε επαφή μαζί του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμά ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να συνομιλούμε απευθεία με τα κράτη-μέλη για πολύ ουσιαστικά νομοθετικά ζητήματα. Και γιατί αυτό, γιατί για την ασφάλεια η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ νομοθετεί τακτικά και συμμετέχουμε σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασία. Πρόσφατα ε, συμμετείχαμε και στο θέμα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία θα ακούσουμε εντός ολίγου που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θέλουμε να ακούσουμε και απευθεία την άποψη των Υπουργών. Και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και τη διαλειτουργικότητα, το ΕΤΙΑΣ ε, και πολλά άλλα ε, θέματα που άπτονται τη αρμοδιότητάς μας. Ε, έγιναν λοιπόν συζητήσεις και τώρα θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τους υπουργούς ε, και ε, συμφωνήσαμε ότι καλό είναι να έχουμε και απευθείας επαφή και χαίρομαι που μετά από το Συμβούλιο Υπουργών ε, μπόρεσαν να έρθουν εδώ σήμερα. δεν είναι έκτακτη συνεδρίαση, είναι σειρά μιας σειρά συνεδριάσεων που γίνονται ε, και χαίρομαι που είναι οι Υπουργοί εδώ για να απαντήσουν τι ερωτήσει μα για τα θέματα αυτά. Θα έχετε την επιστολή που έστειλαν οι δύο Υπουργοί στι 23 Φεβρουαρίου, τη λεγόμενη γερμανογαλλική επιστολή για θέματα που αφορούν εμά κατά προτεραιότητα, τα θέματα προτεραιότητα στο διάλογο ασφαλεία. Περιλαμβάνουν βέβαια και πολλέ από τι δικέ μα τι προτεραιότητε, αλλά μπορεί να δίνουμε διαφορετική ε, σημασία στα διάφορα θέματα και επομένω μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε και φαντάζομαι ότι αυτό θα κάνετε. Αλλά ήθελα να σα ζητήσω να επικεντρωθείτε κυρίω στο διάλογο για την ασφάλεια. Ε, είναι βέβαια ανοιχτή η συνεδρίαση για σας. Αν θέλετε να θέσετε άλλες ερωτήσεις ε, στους δύο υπουργούς, ε, το Γάλλο και το Γερμανό Υπουργό, βεβαίως και μπορείτε. Να προχωρήσουμε τώρα στη συζήτηση. Ε, μας πιέζει λίγο χρόνος. Πρέπει να τελειώσουμε γέρος αυτή τη φορά. Θα ήθελα λοιπόν να με βοηθήσετε όλοι. Όταν καθορίζω όρια, ακόμα και για τους υπουργού, θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε τους χρονικούς περιορισμούς. Και θα κάνουμε το εξής. Θα δώσω από ένα τέταρτο στον κάθε υπουργό, αλλά συμφωνήσαμε προηγουμένως πολύ φιλικά μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας να θα συζητήσουμε σε θεματικές ενότητες αυτά τα 15 λεπτά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Φέκολ, ο οποίος θα αναφερθεί για τρία λεπτά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμεζιέρο, ο οποίος θα μιλήσει για τη διαλειτουργικότητα και θα συνεχίσουμε έτσι. Σας καλωσορίζω λοιπόν κύριε Υπουργέ. Και σας παρακαλώ να ξεκινήσετε τη συζήτηση και να μας δώσετε την άποψή σας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Ντεμεζιέρ, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για αυτήν την ακρόαση. Πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής, αλλά αισθάνομαι και ε, μεγάλη τιμή για αυτή την πρόσκληση λίγες μέρες ε, μετά τον ορισμό μου. Ο προκάτοχός μου, ο κ. Σουαλερού, ε, είχε λάβει την δέσμευση να έρθει εδώ και βεβαίως εγώ δεν θα μπορούσα ε, να μην ε, προσυπογράψω τη δέσμευση αυτή πρώτα απ' όλα γιατί εκπροσωπείται το ευρωπαϊκό όνειρο των πολιτών αλλά και εξάλλου γιατί έχω μεγάλο σεβασμό απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις προηγούμενες θέσεις και ευθύνε που είχα πάντα προσπάθησα να συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, εκφράζει την νομιμότητα και την νομιμοποίηση μάλλον τη δημοκρατική στο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και επίση ένα άλλο λόγο ήταν γιατί θα είχα την ευκαιρία να συνεχθούμε με τον κύριο Δημιζιέρ, ε, διότι τρέφω πάντα μεγάλη εκτίμηση στη Γερμανία. Ε, έχετε αυστήρου κανόνε θέση και επομένω θα ξεκινήσω. Όσον αφορά την αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, θα σα πω δύο λόγια σχετικά ε, με την Γαλλία. Γνωρίζετε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο απειλής, πράγμα που επεβεβαιώνει επιβεβαιώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα από το χτύπημα στο Λονδίνο, αλλά και πριν από αυτό ε, στην ε, ε, Ευρώπη είδαμε να πλήττονται πάρα πολλές χώρες από τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις. Επομένως είδαμε μέσω της εδώ στην προκείμενη περίπτωση της Αγγλίας είδαμε να θίγεται άμεσα το σύμβολο της δημοκρατίας, το κοινοβούλιο. Ε, είχαμε επίσης την περίπτωση της Αμβέρσας ε, ε, όπου συνελήφθη ένα άτομο και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρομοκρατικές ενέργειες. Καμία χώρα, κανένας πολίτης δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι προστατευμένος από τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό δυστυχώς είναι το χαρακτηριστικό της της ε, εποχής και θα πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να προστατέψουμε τους πολίτες μας. Μέχρι τώρα μαζί καταφέραμε ε, να ε, πετύχουμε κάποια πράγματα σημαντικά, αλλά ακόμα παραμένει πολλής δρόμος. Γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν σε πολλές περιπτώσεις έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πρώτα απ' όλα γιατί ε, ως προστάτητα των ε, θεσμών και θεματοφύλακα των συνθήκων βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και γιατί ακριβώς εκπροσωπεί ε, την, τον αγώνα των λαών κατά της τρομοκρατίας των πολιτών της Ευρώπης. Ε, εμείς ε, έχουμε ε, προχωρήσει σε λήψη μέτρων καθώς επίσης και τη δημιουργία νέων εργαλείων. Σε αυτά τα πλαίσια και με αυτήν την φιλοδοξία τον Φεβρουάριο του 2017 μαζί με την Γερμανία ο προκάτοχός μου απίφθινε επιστολή σε ευθεία γραμμή με τις αποφάσεις του Ιουλίου του 2016 πρώτη πρώτη πρόκληση, πρώτο επίδικο αντικείμενο είναι ε, η πραγματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στόχος απαραίτητο να επιτευχθεί έτσι ώστε να προστατευτούμε από την τρομοκρατία αλλά ε, και για να είμαστε σε θέση καλύτερα να ταυτοποιήσουμε και επομένως ε, να ελέγξουμε και τις μεταναστευτικές ροές. Είναι απαραίτητο έτσι ώστε να παραμείνει η Ευρώπη χώρος ελευθερίας ε, και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν τα κοινά μα σύνορα ε, είναι ασφαλή, γιατί διαφορετικά το σύνολο του ευρωπαϊκού σχεδίου θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα σα πω και ποια μέτρα έχουμε πάρει. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις ε, ε, επιτύχαμε συμφωνία ε, όσον αφορά ε, την οδηγία βάσει της οποίας καταχωρούνται όλοι οι επιβάτες στο, των αεροπορικών εταιριών, το γνωστό ευρωπαϊκό PNR. Το συζητήσατε πολύ και στο Κοινοβούλιο. Αναθεωρήσαμε επίσης τον κώδικα, τον, τον κώδικα Σέγγεν των συνόρων έτσι ώστε να ε, υπάρξουν σε πολλές περιπτώσεις έλεγχοι ε, για τους πολίτες της Ευρώπης ε, και τους πολίτες των τρίτων χωρών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε ανέπαφο τον εσωτερικό χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας. Επίσης, εγκρίναμε ε, την ε, ε, οδηγία, εγκρίνατε μάλλον εσείς εδώ τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με την έκβαση γιατί η συζήτηση υπήρξε μακρά και περίπλοκη του θέματος αυτού πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να περιορίσουμε την πρόσβαση στα επικίνδυνα όπλα ε, και να περιορίσουμε την ε, πρόσβαση στην πηγή των όπλων. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η χνηλασιμότητα ε, των όπλων. Τα πρώτα μέτρα αυτά αποτελούν πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, θα ακολουθήσουν βεβαίως και άλλα εν ευθέτω χρόνο, αλλά γνωρίζουμε ότι ο καθένας το ρόλο του με τις απαιτήσει του και τις προϋποθέσεις του, μπορεί να έχει μαζί σας έναν αυστηρό και απαιτητικό διάλογο. Μπορεί σε εσά ε, να βρει έναν ε, αυστηρό ελεγκτή, ε, ο οποίος όμως βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά ήθελα να σας πω για τα πρώτα τρία μου λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. τώρα θα σας ε, θα, δώσω το λόγο στον κύριο Ντεμεζιέρ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι. Η κυρία Ζήπελ από τη Γερμανία μας καλωσήρισε πριν από λίγο και μας είπε ότι αν κοιτάξουμε τις ε, επωνυμίες, τα ονόματα, ο Γάλλος Υπουργό έχει γερμανικό όνομα και ο Γερμανός έχει γαλλικό όνομα. Σύμπτωση, μεν, σημαδιακή ιδέα. Ξέρετε ότι η Γαλλία και η Γερμανία σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια βρουν από κοινού. από τότε που ήταν ο Μπερνάρ Καρνόφ ε, υπουργό εσωτερικών και από πριν και από τότε που ήμουν και εγώ ε, υπουργό. Ε, και θέλουμε ασφαλώς να συνεχίσουμε την παράδοση αυτή. Τρέφουμε μεγάλη σεβασμό για την εργασία της Επιτροπής αυτής και ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, μεν διαφορετικές απόψεις, αλλά νομίζω ότι από το PNR έχει καταστεί τουλάχιστον ε, σαφές ότι ε, μπορούμε, δεν είμαστε αντίθετοι και αντίπαλοι, να συνεργαζόμαστε. Μπορούμε λοιπόν να Δεν μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε τι διαπραγματεύσεις τόσο, μακροπρο... τόσο μακρόχρονες όπως για το PNR. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και από κοινού του με τον Γάλλο συναδελφό αδελφό μου θα ήθελα να απευθύνω και εγώ έκκληση για μια γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία. Αυτό που συμβαίνει συχνά με τι ε, οδηγίε και του οικονομισμού, εγώ θα ήθελα μάλλον να μην μιλήσω καμία οδηγία, να μιλήσω για μια αρχή, για την αρχή της διαλειτουργικότητας, για καλούς λόγους και για βάσιμους λόγους ε, κατά το παρελθόν. Τα ζυγίσαμε όλα και αποφασίσαμε για διάφορους σκοπούς να δημιουργούνται διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές, διαφορετικοί κανονισμοί. Αυτό το Eurodact, το Schengen, ε, Information System, Prune και πολλά άλλα τέτοια συστήματα. Η Eurodact λοιπόν ε, έχει αντακτικά αποτυπώματα και χωρίς ονόματα. Το Schengen, το SIS ε, έχει ονόματα, δεν έχει αντακτικά αποτυπώματα. Και όταν έγιναν τα μεγάλα χτυπήματα στην Γαλλία, είπαμε και εμείς και εσείς ότι δεν είναι δυνατόν ε, οι υπηρεσίες ασφαλείας να μην έχουν πληροφορίες τις οποίες έχουν άλλες ε, αρχές. Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή απόψε ε, δεδομένων. Τίθεται και νομικά ζητήματα αλλά και τεχνικά ζητήματα, ουσιώδη. Στο Συμβούλιο υπάρχει λοιπόν πλέον μια ομάδα υψηλού επίπεδου πλέον η οποία καταθέτει σχετικές προτάσεις για το θέμα αυτό και θέλουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του ΣΥΣ και τη Eurodac. Δεν θέλουμε λοιπόν να περιμένουμε μέχρι ότου επιληφθεί το θέμα της διαλειτουργικότητας. Αλλά αποτελεί ένα βασικό ζήτημα. Και όσοι προσπίζονται τα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να πω το εξή. Υπάρχει αυτή η έννοια της λιτότητας των δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν αυτή η αρχή και ισχύει για πολλά δεδομένα. Αλλά μπορούμε να κατανοήσουμε και με διαφορετικό τρόπο αυτή τη λιτότητα δεδομένων, ότι καταγράφουμε και αποθηκεύουμε μόνο μία φορά τα δεδομένα. Και οι αρχές θα πρέπει να φροντίσουν να ανταλλάσσονται τα δεδομένα αυτά και να υπάρχει και ένα έξυπνο σύστημα πρόσβασης για να υπάρχει πρωτοκόλληση και προκειμένου να υπάρχει σωστή και καταγεγραμμένη πρόσβαση στα δεδομένα θα μπορούσαμε ενδεχομένω να αποφύγουμε και τη συλλογή κάποιων δεδομένων. Αν ε, μπορούσαμε να συνδυάσουμε κάποια δεδομένα τα οποία ήδη υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το θέμα τη διαλειτουργικότητα. Προ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε και θα χαιρόμουν ιδιαίτερω αν ακολουθήσετε και εσεί αυτή την οδό. Ο πρόεδρο. Δεν ξέρω τι δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλία και Γερμανία, αλλά ήταν πιο κοντά στο όριο που σα έδωσα η ομιλία σα, η παρέμβασή σα. Ευχαριστούμε λοιπόν, Τόμα. Και αν αναρωτιέστε γιατί εξετάζουμε κάθε μεμονωμένο τομέα, γιατί ναι μεν θέσαμε ε, μια τακτική με την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε κάποια βασικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, το θέμα της τεχνολογίας, φυσικά το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έτσι οδηγούμαστε στα ζητήματα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Ε, ε, Ο κ. Φέκλου θα αναφερθεί στο ETA, στο Eurodac και στα λοιπά. Έλαβα το έμαθα για το χρόνο μήνυμα ελήφθη. Είναι απαραίτητο ναι, αυτό το οποίο ακούστηκε. Η διαλειτουργικότητα είναι σημαντική γιατί τα συστήματα λειτουργούν καλά και επομένω για τον εξή απλό λόγο. Παντού στην Ευρώπη κάθε υπηρεσία ασφαλεία θα πρέπει να μπορεί σε πραγματικό και σίγουρα σε χρήσιμο χρόνο να έχει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε προκειμένου να γνωρίζει ε, με ποιον έχει να κάνει και κυρίω αν υπάρχουν χρήσιμε πληροφορίε για το συγκεκριμένο άτομο. Γι' αυτό λοιπόν στην αρχή ήμασταν υπέρ τη δημιουργία ενό ενός σύστημα τόσο εισόδου-εξόδου και πάλι με τη λογική να ε, έχουμε ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα. Χαιρόμαστε που προχωρούν τα πράγματα από αυτού, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει σε αυτές τις εργασίες να συμπεριλεύουμε και ε, κοινοτικούς ε, ε, πολλά έγιναν από Ευρωπαίους πολίτες. Επομένως πρέπει να γνωρίζουμε εάν έφυγαν, γύρισαν, αν πήγαν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ε, τις μετακινήσεις τους. Βεβαίως ε, γι' αυτό σεβόμαστε την αρχή της ε, αναλογικότητας και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρά, ξέρω ότι τα προσέχετε αυτά, ε, αναλογικότητα για να σεβαστούμε και την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και αυτά τα δύο δεν ε, είναι αντίθετα μεταξύ των, δεν είναι ανταγωνιστικά. Ε, λαμβάνονται όλες οι εγγύησει για την πρόσβαση και τη διατήρηση αυτών των δεδομένων και μόνο τα απαραίτητα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν και θα ε, τα διαβουλεύονται οι αρμόδιοι. Ε, το ΕΤΙΑΣ όσον αφορά τα ταξίδια στο οποίο αναφερθήκατε ε, θα λειτουργήσει και θα είναι γρήγορα αποτελεσματικό. Θα μπορούμε να δούμε ε, ποιοι ε, υπόκοοι τρίτων χωρών έχουν απαλλαγή θεώρησης διαβατηρίων, κατά πόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να βρεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την άφηξή τους και ε, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν αποτελούν απειλή ε, για το κοινωνικό σύνολο. Επίσης ε, θέλουμε να δούμε κατά πόσον οι υπηρεσίες καταστολής και οι συνοριοφύλακες σε όλα τα κράτη-μέλη έχουν ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση στα σύστημα ε, στη σύμμετα πληροφοριών θεωρήσεων διαβατηρίων και στην βάση Eurodac. Ε, σας, ε, μου περίσσεψε και λίγο χρόνος, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθείτε να κερδίσετε πιστώσεις εδώ χρόνου για να σας δώσουμε μετά. Παίζετε παιχνιδάκια, αλλά καλό είναι αυτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ να σας πω ότι μετά από τρεις ημέρες ε, δεν θα ήμουν σε θέση να παρέμβω και πραγματικά τα σέβομαι προς τον Ματίας. Ε, να πω δύο πράγματα για το Exit ε, Entry System, γιατί έχει να κάνει και αυτό με το SIS, Schengen Information System. Ε, θέλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθεσία αυτή μέχρι τα τέλη του χρόνου. Βρισκόμαστε σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σύστημα εισόδου-εξόδου θεωρώ ότι αποτελεί για μένα την κατεξοχήν βασική προϋπόθεση για την συνεχίση ελέγχων συνήνωρων για το Σέγγεν, για τον χώρο Σέγγεν. Χωρίς ε, σωστό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων δεν θα υπάρχει στο μέλλον πραγματικά πραγματικός χώρος, ιστορικός χώρος Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο κέρια σημασία. Γι' αυτό λοιπόν το σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν για, την ασφάλεια, για τις υπηρεσίες ασφάλειας μάλλον είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο, με μεγάλη χρονοκαθυστέρηση βέβαια, ε, δημιουργήθηκε και με μεγάλη αύξηση του κόστους και με πολύ πολύ πολύ ενόχληση. Αυτά έχουμε παρατηρήσει ως τώρα. Στη συνέχεια, μετά τις επιθέσεις στη Γαλλία, προσπαθήσαμε να βάλουμε στο σύστημα πληροφόρηση Schengen για τους foreign fighters, για τους αλλαδαπούς ε, μαχητές ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραμποδίσουμε, να μην παρακολουθήσουμε το σύστημα. Πλέον όμως διαπιστώσαμε ότι δεν αρκεί αυτή η ένταξη και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν νέες κατηγορίες ε, ε για διαγωνισμούς με νέα βιομετρικά στοιχεία, με ε, δεσμευτικούς όρους σε ό,τι αφορά τους τρομοκράτες ε, και σε ό,τι αφορά επίσης επέκταση των δικαιωμάτων πρόσβασης και για τις φορολογικές ε, υπηρεσίες και για τις μυστικές υπηρεσίες και το καθεξής. Πολλά από αυτά ήταν αφιλεγόμενα και ε, προσβλέπουμε στη συζήτηση μαζί σας των βασικών αυτών ζητημάτων. Ωραία, τώρα θα μιλήσετε εσείς ε, κύριε Φλάκη για τις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Ε, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ε, κρυπτογράφησης και ο τρόπος με τον οποίο ε, συνεργαζόμαστε με τους φορείς του διαδικτύου για την αποκρυπτογράφηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το, η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική για την τρομοκρατία. Ε, εμείς έχουμε πολλούς operators απέναντί μας οι οποίοι δεν είναι πολύ συνεργάσιμοι ε, ε, ε, έχουμε αυτή τη στιγμή δυστυχώς μια κατάσταση η οποία δεν μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση de facto σε περιεχόμενο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα νομικό εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να υποχρεώνει έναν πάροχο να συνεργαστεί με τις αρχές. Γι' αυτό λοιπόν από κοινού η Γερμανία και η Γαλλία έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο ε, να υποβάλει ε, τους ε, παρόχους περιεχομένου διαδικτύου στις ίδιες υποχρεώσεις που υποβάλλονται οι παροχή τηλεφωνίας. Ήδη αναφέρθηκε από τους Βρετανούς συναδέλφους μας και ομολόγους μας ότι μέσω του WhatsApp αυτής της εφαρμογής βοηθήθηκε η τρομοκρατική ε, ε, το, το τρομοκρατικό πλήγμα στο Westminster. Θέλουμε να σας διασφαλίσουμε ότι είναι απαραίτητο βεβαίως να διατηρηθεί το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες ε, στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν συστήματα ε, ιδιαίτερα αυστηρά τα οποία ταυτοχρόνως επιτρέπουν την ελευθερία των πολιτών και την προστασία της ιδιωτικής του ζωής αλλά και την προστασία της ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές ε, οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει όλη η Ευρωπαϊκή ήπειρο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, πάντα σεβόμενη το δίκαιο. Ευχαριστώ. Και μια μικρή παρατήρηση για γι' αυτό μου επιτρέπετε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ε, τηλεμέσων έχουμε ε, ενημερώσει ε, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παρακολουθούμε τηλέφωνα με τηλέφωνα και ε, τα τηλεμέσα ακολουθούν τους κανόνες των τηλεμέσων. Λειτουργικά όμως αυτά εξελίσσονται από κοινού. Είτε μιλάμε για το σταθερό δίκτυο, είτε μιλάμε για τα smartphones, είτε για τα voice over IP, είτε τηλεφωνούμε μέσω Skype, λειτουργικά το ίδιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά η νομοθεσία είναι εντελώ διαφορετική. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Άρα από τεχνική ε, πλευρά, από τεχνική καταταξή τη νομοθεσία, θα πρέπει να περάσουμε σε μια λειτουργική ε, κατάταξη και τα τηλεμέσα και τις τηλεπικοινωνίες να τα βάλουμε σε ένα καλάθι. Και αυτό α, κατά το δυνατόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξουν εθνικοί κανονισμοί. Και αυτό θα δημιουργήσει σε κατακριματισμό και προβλήματα. Αυτό είναι, που είναι σημαντικό είναι η αρχή ε, του τόπου αγοράς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τις χώρες ε, της Ευρώπης και κάτι που ανέφερε και ο Ματίας. Το ζήτημα της ε, διασύνδεσης. Και εδώ να προσπαθήσω να διευκρινίσω μία παρανόηση. Χρειαζόμαστε κωδικοποίηση στο διαδικτύο για να υπάρχει ασφάλεια και χρειαζόμαστε επίσης ασφάλεια παρά την ε, κωδικοποίηση. Είμαστε λοιπόν end-to-end end to end κωδικοποίηση. Θέλουμε και οι ιδιώτε να έχουν ε, κωδικοποίηση, δεν θέλουμε backdoors, αλλά αντίστροφα δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίε ασφαλεία, μόνο με κάποια μέσα να μπορούν να αποφεύγουν ε, ποινική δίωξη. Δηλαδή, οι υπηρεσίε ασφάλεια ε, δεν χρειάζονται να έχουν πιο, πολύ, ή πιο πολλά ή πιο λίγα δικαιώματα από ότι διαδικτύου. Άρα το θέμα της ε, κωδικοποίησης end-to-end είναι πολύ σημαντικό και θα είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Έχουμε το θέμα της επικοινωνίας πηγής ε, στο διαδίκτυο. Όλα αυτά είναι τεχνικός πώς πάρα πολύ περιπλόκα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Γαλλία. Αυτή ήταν λοιπόν η διπλή μας παρουσίαση κύριε Πρόεδρε και φυσικά σήμερα Έχουμε σήμερα πάρα πολλά να συζητήσουμε για το relocation resettlement, για την μετανάστευση, αλλά το θέμα σήμερα λοιπόν είναι η τρομοκρατία και η ασφάλεια. Και δυστυχώ παρά τις, ε, το γεγονό ότι μέχρι τι 7 θα λάβει η χώρα η σημερινή συνάντηση, εγώ θα πρέπει να φύγω στι 7 παρατέταρτο για να προλάβω το αεροπλάνο μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Um, Νομίζω ότι όπως διοργανωτική συζήτηση δεικνύει ότι ότι ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική η παρουσίασή σας. Σημειώνω ότι θα πρέπει να φύγετε λίγο πιο νωρί. Γι' αυτό λοιπόν να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συζήτηση. Και επειδή θέλετε να υπάρξει και κάποια feedback από τον Τόμας Δεμαζιέρ, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά. Και να πάμε κατευθείαν στους ομιλητές. Όποιοι δεν έχουν ζητήσει το λόγο παρακαλώ τώρα να το ζητήσουν και πώς θα, διοργανωθ... πώς θα δώσουμε απαντήσεις. Κατευθείαν. Κοιτάξτε. Να σας ακούσουμε εσάς πρώτον. Και αν είσαστε όλοι παρακαλώ, θα τηρήσετε τα χρονικά όρια. Όποιοι δεν έχουν ζητήσει ακόμα το λόγο, παρακαλώ να το ζητήσουν τώρα. Σήκωστε τα χέρια σας. Ξέρω ότι είναι λίγο σαν να στο σχολείο, αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Να κλείσουμε το κατάλογο. Ξεκινάμε με τους συντονιστές. Κανένας πάνω από δύο λεπτά σας παρακαλώ. Η κυρία Μέτσολα πρώτα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους Υπουργούς ε, Φέκλου και Τεμεσγέρ που είναι εδώ σήμερα. Συμφωνώ απολύτως και με τους δυο σας όταν λέτε ότι μόνο μέσω της εξασφάλισης των εξωτερικών συνόρων θα μπορέσουμε να απολαμβάνουμε τις ελευθερίες που μας προσφέρονται ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα εντός αυτών των ε, συνόρων. Και όταν αναφερόμαστε στη διαλειτουργικότητα και πλήρη ανταραγή πληροφοριών, είναι πάρα πολύ σημαντικό μεν αυτό, αλλά ταυτόχρονα ορισμένε φορέ είμαστε και πάρα πολύ αργοί στην έγκριση νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλά χρόνια μετά την ανάγκη για αυτή την νομοθεσία ε, και η ερώτησή μου θα είναι σύντομη. Όταν αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως είπατε και εσείς, είναι παγκόσμια μάχη και επομένω χρειάζεται και παγκόσμια απάντηση. Αν εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, Πώς ε, βλέπετε να προχωράει αυτή η σχέση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη απάντηση από αυτή που είχαμε μέχρι τούδε, βάσει και των κοινών αξιών των δύο υπήρων για την αντιμετώπιση της απειλής και ε, μετά. Στη συνέχεια των επιθέσεων του Βερολίνου τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε μια συζήτηση με τον Επίτροπο Κίνγκ ε, την περασμένη εβδομάδα και διαπιστώθηκε ότι οι τρομοκράτες ε, που έκαναν τις επιθέσεις είχαν χρησιμοποιήσει 14 διαφορετικές ταυτότητες. πέρα από τη νομοθεσία που έχουμε στα σκαριά ε, τι κάνουν οι χώρες σας ε, για να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τα βιομετρικά δεδομένα. Υπάρχουν εξελίξεις πέραν ε, των νομοσχεδίων και την αξιολόγησή τους αυτή τη στιγμή στη συνεργασία που μας παρουσιάσατε τόσο εύγλωτα εδώ. Ευχαριστώ η Birgit για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία μικρή παρατήρηση, επιτρέψτε μου. Ο Γερμανός υπουργό είπατε έχει γαλλικό όνομα και αντίστροφα. Ο Γάλλος υπουργό είναι γερμανικό. Εγώ δεν σκέφτομαι τόσο πολύ τι γαλλογερμανικέ σχέσει, να σα πω την αλήθεια. Εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι κάποιε περίεργε συζητήσει που γίνονται στην Ευρώπη για την διατήρηση τη εθνική ταυτότητα. Για μένα αυτά τα δύο ονόματα ξεκαθαρίζουν ότι όχι μόνο στη Γαλλία και στη Γερμανία, αλλά παντού στην Ευρώπη είναι... Είμαστε μεικτοί, ανάμεικτοι, γιατί η μετανάστευση των προηγούμενων αιώνων νομίζω ότι έχει αναμίξει όλες μας τις χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ως ε, παρατηρήσει, να θέσω το θέμα της, ε, του διαλόγου για, τον, ε, για την ασφάλεια, το θέμα της διαλειτουργικότητας. Θα σας προκαλέσει ενδεχομένε έκπληξη το γεγονός ότι μπορώ να συμφωνήσω με διάφορα από αυτά που είπε ο Υπουργός του Μέιζερ. Αλλά αν θέλουμε να υπάρξει διαλειτουργικότητα, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Καταρχάς, ποιος θα έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα. Αυτό δεν απασχολεί μόνο τους ε, ακτιβιστές και αυτούς που θέλουν να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά όλες τις αρχές, τις αστυνομίες, τις υπηρεσίες ασφάλειας, ε, δεν μπορούν όλοι ε, ενδεχομένω να έχουν την ίδια πρόσβαση στα δεδομένα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο και το ακούσαμε ότι χρειαζόμαστε ενιαίους ορισμούς ποιος είναι, από πότε, από ποια στιγμή τρομοκράτης, ποια είναι η στιγμή που θεωρείται ύποπτος. Γιατί φυσικά αν δεν υπάρχουν ενιαίοι ορισμοί είναι αδύνατο να υπάρξει ασφάλεια των δεδομένων. Ένα άλλο θέμα, η χρήση των δεδομένων ε, του συστήματος ΣΥΣ, του Eurodac. Θα ήθελα να εκτιμήσουν, να ακούσουμε την εκτίμηση των Υπουργών στο σημείο αυτό, γιατί στις πρώτες επιθέσεις εδώ στο Βέλγιο είχαμε την εντύπωση ότι οι βάσεις δεδομένων όπως ε, το ΣΥΣ δεν χρησιμοποιούνται εγκαίρως. Είναι τεχνικό μόνο το ζήτημα. Ήθελα να ξέρω. Και τελευταίο για την ε, κρυπτογράφηση. Είναι δύσκολο το θέμα, γιατί αν έχω κάποια υποψία μπορώ να ανοίξω μια επιστολή σε ό,τι αφορά την κρυπτογράφηση. Μπορώ να αναπτύξω μια τεχνολογία για να διαβάσω ένα mail ή χρειάζεται ένα γενικό κλειδί. Και υπάρχει σε την περίπτωση αυτή η δυνατότητα να εμπιστευτούμε τις αρχές μας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και του ε, εμπειρογνώμονες και του υπουργού επ' αυτού. Συνάδελφοι, προσπαθήστε να τηρήσετε τα δύο λεπτά και μην νομίζετε ότι πρέπει να τα πείτε όλα σε δύο λεπτά. Τα καλύπτετε όλα μένα, αλλά προσπαθήστε να καλύψετε τα ουσιώδη. Η Χέλγα Στίβεν για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, δύο υπουργού για την παρουσίαση και χαίρομαι και εγώ με την πρότασή σας για να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ αφενός της ασφάλειας και αφετέρου της ιδιωτικής σφαίρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Παρίσι και τις Βρυξέλλες έλαβε πολλά συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσει την ασφάλεια για τους πολίτες μας. Διάφορα μέτρα όπως για παράδειγμα ο έλεγχος των διεθνών μεταφορών και ε, έλεγχος των Ευρωπαίων υπηκών ε, είναι, έχουν δρομολογηθεί. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία για τις εθνικές ε, κυβερνήσεις. Αλλά τι προληπτικά μέτρα, μάλλον λοιπόν πολλά προληπτικά μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόληψη της ε, τρομοκρατίας. Για παράδειγμα, στον Πόλεμπέικ δραστηριοποιούνται 51 τρομοκρατικές διγαντιστικές οργανώσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Το Βέλγιο ξεκίνησε μόλις με τον έλεγχο των μεταφορών με λεωφορείο πέρα από των ε, τρένων. βλέπετε τέτοια ε, μέτρα PNR σύντομα και πότε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιντφέλτ από τους φιλελεύθερους. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Πολλά μπορούμε να πούμε για όλες τις προτάσεις, αλλά και για τις διαδικασίες. Αυτό είναι ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τα πιο ενοχλητικά. Σε μια δημοκρατική κοινωνία πιστεύω ότι η νομοθεσία, ιδίω η νομοθεσία που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων, πρέπει να εγκρίνεται με τον πιο διάφανο τρόπο και είναι πολύ ωραίο που κάθεστε και σχεδιάζετε από κοινού. Έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να συζητηθεί στο Συνοβούλιο, στο Κοινοβούλιο ε, και να περιμένετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις. Καλύτερα αυτό. Και πρέπει να πω ότι ανησυχώ για νέες προτάσεις όταν ακούμε ότι οι προτάσεις οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί δεν εφαρμόζονται. Έγιναν αρκετέ ανταλλαγέ απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό PNR, τα στοιχεία των ε, πτήσεων των επιβατών. Ε, ε, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, μα πιέζεται για να περάσει γρήγορα αυτή η νομοθεσία. Έχει περάσει ένα χρόνο μετά την ψηφοφορία και τι έχει γίνει. Από ό,τι γνωρίζουμε μόνο ένα κρατός έχει κάνει πλήρη εφαρμογή και αυτό ήταν και πριν από την έγκριση και όλοι οι υπόλοιποι απλώ ενδιαφέρονται. Πού πήγε αυτό ο κατεπήγον χαρακτήρα. Και επίση γνωρίζουμε ότι μετά από κάθε επίθεση διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπήρχαν πληροφορίε διαθέσιμε στι υπηρεσίε, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν κατά και στην επίθεση, περίπτωση επίθεση του Βερολίνου κρίνω. Υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ε, προηγουμένως από την αστυνομία της Γερμανίας που έλεγε στις αρχές ότι είναι επικίνδυνο ο συγκεκριμένο άνθρωπος. Αλλά τελικά δεν έτυχε της κατάλληλης αξιολόγησης και δεν ήταν υποκράτης αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, κάθε φορά που γίνεται επίθεση, σαν την επίθεση στο Westminster την προηγούμενη εβδομάδα, είναι φρικτό το γεγονός, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τι είναι τρομοκρατία. Γιατί η αίσθηση που έχω εγώ από τις εφημερίδες, και δεν είμαι και αστυνομικός, πρέπει να βασιστώ στα όσα διαβάζω στα μέσα, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ε, υπό την επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, είναι τρομοκράτης ακριβώς αυτός. Ε, και τέλος, μια τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε προσπαθούμε να εξεύρουμε τη δέουσα ισορροπία και έχουν και δικαίωμα οι πολίτες ε, να ζητούν ε, ε, να δικαιωθούν για την πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, ε, ε, πρόσβαση σε εμπιστευτικά δικαιώματα. Αναφέρομαι και στο δικαίωμα ε, να δικαιωθεί κάποιος στη Γαλλία, το αναφέρομαι σε εσά κύριε Υπουργέ, και αν θέλουμε να έχουμε περισσότερες εξουσίες για τις αρχές, πρέπει να έχουμε και περισσότερες δικλείδες ασταλίας για τους πολίτες και εκεί υστερούμε πάρα πολλές τις προτάσεις μας. Το ξέρω ότι ότι μια και είναι εδώ οι Υπουργοί θέλετε να αναφέρετε όλα τα προβλήματα, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό. Λίλια Ένστα από την Κούα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να καλωσορίσω και τους δύο υπουργούς εσωτερικών από την πλευρά τη ομάδας μα. Έχω τι εξής ερωτήσεις, ε, κοιτώντα τι πρόσφατε επιθέσει ε, στο Βερολίνο, στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, στο Λονδίνο και στι δύο περιπτώσει. Το PNR δεν θα έχει χρησιμεύσει σε τίποτα μας ε, διακηρύτεται ότι το PNR ε, μας χρειάζεται για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, ότι στο Βέλγιο οι επιθέσεις που έγιναν είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί οι τρομοκράτες και στο Παρίσι και το 2010 στο Λονδίνο. Ε, αυτοί που έκαναν τις επιθέσεις ήταν γνωστοί ως τρομοκράτες. Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετική η προσέγγιση και όχι απλά να συλλέγουμε όλο και πιο πολλά δεδομένα, αλλά αντικειμενικά να εξετάζουμε τι μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για ενδεχόμενους ε, για ενδεχόμενα άτομα που θα κάνουν επιθέσεις ε, και να υπάρχει καλύτερες ε, δικτύωση μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών, μεταξύ κρατών μελών, αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Εκεί να εστιαστούμε. Το, κατά δεύτερον, η αρχή της τρομοκρατίας. Δεν μας πει καθόλου ο όρος αυτό σε ό,τι αφορά το εύρος εφαρμογής τους και είναι όλο και πιο δύσκολο να, να καθοριστεί το τι αποτελεί τρομοκρατία και τι όχι. Γιατί αυτό προφανώς έχει να κάνει και μια, μια ομάδα δεδομένων. Τρίτο σημείο προς τον Γάλλο συνάδελφο. Μιλήσατε και έχετε μέχρι τον Ιούλιο 2017 έχετε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι σας αποφέρει αυτό, μήπως θα πρέπει επιτέλους να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τα μέτρα για την καταπολέμηση της, δημο... της τρομοκρατίας και το καθεστώς πραγματικά εκτάκτης ανάγκης για τέτοιο μακροχρόνιο διάστημα έχει αποτελέσματα, το έχετε εκτιμήσει αυτό. Και τελευταίο, η κρυπτογράφηση, εδώ θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εγώ δεν έχω οποιαδήποτε διάθεση να κάνω οτιδήποτε εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι εγκυμονεί πολλούς κινδύνους το μέτρο αυτό. Ο Πρόεδρος. Για τους πράσινους η κυρία Σκά Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα ρωτήσω πράγματα για την ασφάλεια. Ε, αναρωτιέμαι τι γίνεται με την relocation. Ε, έχετε και οι δύο τέτοια ε, σχέδια. Κύριε Ντεμεζιέρε, εσείς ε, προσπαθήσατε να προωθήσετε το θέμα του και τα προγράμματα relocation, αλλά νομίζω ότι από την Ελλάδα και από την Ιταλία δεν έχουν μετακινηθεί πάρα πολύ και φαίνεται ότι η Γαλλία έχει καλύψει 14% από την ποσόστοση, η Γερμανία 11% και αυτό από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο φαντάζεστε ότι μπορεί να ε, εντατικοποιηθεί ε, η διαδικασία relocation από αυτές τις συγκεκριμένες χώρες. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε ε, με άλλες χώρες γιατί βλέπουμε ότι η Αυστρία προσπαθεί να βγει από το πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει τι θα κάνετε έτσι ώστε να ξεφύγουν οι άνθρωποι αυτοί από αυτές τις φρικτές συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Καταλαβαίνω ότι ε, μάλιστα εσείς οι δύο προετοιμάζεστε να επιστρέψετε στην Ελλάδα κάποιους ε, ε πρόσφυγες. Σω εάν, τώρα θα δώσω το λόγο σε εσά, εάν είσαστε σύντομοι, ενδεχομένω θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και άλλε ερωτήσει. Η κυρία Χολμάιερ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί Υπουργοί, που βρίσκεστε εδώ πέρα στην Επιτροπή μαζί μα. Έχω τι εξή ερωτήσει. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με την αξιοποίηση των δεδομένων, τη τραπεζών των δεδομένων και σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων από κράτη-μέλη και σε ό,τι αφορά και την υλοποίηση των ε, νομοθεσιών. Αναρωτιέμαι, στο σύστημα PNR έχουμε 28 εθνικά συστήματα, γιατί δεν υπήρχε μετά διαμορφώσεις σε ένα ευρωπαϊκό συστήματος. Μπορούμε να έχουμε μια εγγύηση ότι εξ αρχής θα ληφθεί υπόψη η διαλειτουργικότητα και θα λειτουργήσει 100% σε ό,τι αφορά και τις επιθέσεις του Μπατακλάν, σε ό,τι αφορά την Αλκάιντα, ότι μπορούν να α, υπάρχει μεταφορά σε όλη την Ευρώπη για το ποιο έφυγε από το Παρίσι, ποιο πήγε στη Βιέννη, ποιο πήγε στην Τουρκία. Θα ήταν σημαντικό και τα 28 συστήματα να μην λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, να μην είναι μόνο η πτήση που θα φύγει από τη Γαλλία, αλλά και η πτήση από τη Βιέννη η οποία θα καταγράφεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδη ζήτημα για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε. Και για το Eurodac. Υπάρχει διαρκώ ο φόβο ότι θα ανοίξει για τι ποινικέ αρχέ το Eurodac. Και αυτό θα αποτελέσει γενική υποψία κατά των προσφύγων. Λάμβαναμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτή χρειάζεται και θεωρείται σκόπιμη αυτή η πρόσβαση για προληπτικούς σκόπους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπονιφόη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που είσαστε εδώ και σε ευχαριστώ αγαπητέ Ματιάς ε, που τήρησε σε την υπόσχεση που είχε δώσει ε, ο προηγούμενος ε, προκατοχός σου. Θα ήθελα να επανέλθω στις δύο επιστολές τις οποίες στείλατε δίσε σε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Υπουργή των χωρών σας. Για ποιο λόγο απευθύνεστε στο, στην Κομισιόν και όχι στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως το Συμβούλιο Συμβούλιο υπάρχουν δυσκολίες ε, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμονισμένη κοινή εργασία ε, και ε, επομένως βλέπουμε εδώ ενισχυμένη συνεργασία των δύο χωρών Γαλλίας-Γερμανίας με την Κομισιόν και θέλω και κάτι άλλο να σας ρωτήσω όσον αφορά ε, τους και τους... και την ακτοφυλακή. Ε, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες αναθέσεις που σε μερικές περιπτώσεις μας προβληματίζουν. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό. Δεύτερον, η εναρμόνιση της κατάρτισης ε, που ε, πρέπει να έχουν ε, το προσωπικό ασφαλείας και αστυνόμευσης στα διεθνή τρένα, δηλαδή τα τρένα τα οποία ξεκινούν από το Βέλγιο και πάνε στη Γαλλία κτλ. Πώς βλέπετε τα μέτρα ασφαλείας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο εναρμονισμένα και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε ε, με ποιο τρόπο θα γίνεται η κατάρτιση των ανθρώπων αυτών και σαφώς δεν συμφωνούμε με την πρόταση που υπέβαλε το Βέλγιο να υπάρξει PNR και για τους ταξιδιώτες του τρένου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mrs. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Wickstrom. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργή που ήρθατε σήμερα εδώ ε, ε, και σας ευχαριστώ δε ιδιαίτερο σε εσάς ε, κύριε Ντεμεζιέρα που οργανώσαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση στο Βερολίνο και με δεχτήκατε στο γραφείο σας. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, στο θέμα της μετανάστευσης που είναι σχετικό με αυτά που συζητούμε. Βεβαίως δεν πρέπει να ταυτίζουμε ε, τους μετανάστες ε, με θέματα ασφάλειας, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ξαναβρούμε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αναλάβουν τα θέματα της ασφάλειας σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, αλλά και να ανακτήσουν πλήρως τον έλεγχο ε, τον ε, του, του εσωτερικού χώρου. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξαναβρούμε το σύστημα της μετανάστευσης, την συμφωνία για το άσυλο, το Δουβλίνο, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να περιορίσουμε την πίεση που δέχονται ε, οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και βεβαίως να μειωθεί ταυτόχρονα και ο κίνδυνος ασφάλειας και ταυτοχρόνως όμως να διατηρήσουμε τον ελεύθερο χώρο κυκλοφορίας Σέγγεν που αυτή τη στιγμή δυναμητίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Ντεπρέ, φεύγετε. Καθίστε αμέσως ξανά και πάρτε και το λόγο. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ε, ζητώ συγγνώμη και από τους δύο υπουργού, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να είμαι κάπου στις έξι. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να σας συγχαρώ για αυτή την παρτιτούρα με τέσσερα χέρια που παίξατε. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε τέτοιες ε, καταστάσεις. Ερωτήσεις τώρα. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα καθώς επίσης να υπάρξει και ένα μητρό ε, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να ε, βρίσκει τις πλαστογραφημένες ε, ταυτότητες, πλαστογραφημένα έγγραφα. Μπορείτε να πιέσετε έτσι ώστε να βρούμε αυτά τα κοινά στοιχεία ταυτοποίησης, δηλαδή αυτά τα βιομετρικά στοιχεία τα οποία θα βρίσκονται σε όλες τις ταυτότητες των χωρών. Όσον αφορά το θέμα Σέγγεν, τα έχουμε συζητήσει, αλλά πιστεύω ότι ε, ε, σε κάθε περίπτωση ε, προειδοποίηση στο σύστημα ΣΥΣΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει απευθείας και στο σύστημα καταπολέμησης της τρομοκρατίας της Interpol. Γιατί τι να, γιατί να κάνουμε συστήματα δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Τρίτον, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέτρα για την αποκρυπτογράφηση, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχει τώρα μία τεχνολογία η οποία ονομάζεται CGN και η οποία δίνει την δυνατότητα ή στους providers, ε, στους παρόχους ε, να δώσουν το ίδιο ε, αριθμό IP σε πολλές σε πολλούς χρήστες. Είναι μια τεχνική την οποία έχω επιβεβαιώσει, την έχουν επιβεβαιώσει και οι επαγγελματίες και έτσι γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η ταυτοποίηση. λοιπόν, μαζί με τις τεχνικές αποκρυπτογράφησης, μήπως θα πρέπει να μελετήσετε και και αυτό το θέμα γιατί, ε, τέτοιου, γιατί πολλές έρευνες, πολλές διαδικασίες ε, φτάνουν σε σημεία εμπλοκής ε, σαν αυτά που ανέφερα προηγουμένως και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόνη. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για τα σαφή σας μηνύματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας αυτό, διότι η ουσία είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να σκεφτούμε πώς ε, θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στις διαδικασίες αυτά. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Δύο παρατηρήσει. Πρώτον, η διαλειτουργικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε και τη νέα τεχνική αρχιτεκτονική δομή. Διότι υπάρχουν νέε τεχνικέ δυνατότητε ε, για να υπάρχει πραγματική διαλειτουργικότητα και να ε, προσφέρουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε πληροφορίε σε πραγματικό χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γίνονται αυτά σε πραγματικό χρόνο. Γιατί έτσι επιτρέπεται να δρουν πιο γρήγορα κάποιε αρχέ. Ε, το δεύτερο αφορά τα θέματα ασφαλείας και προστασίας της ιδιωτικότητας, υποχρεώσεις των ε, τηλεπικοινωνιών αλλά και το WhatsApp ε, και ε, διάφορες άλλες τέτοιες υπηρεσίες. Ξεκινάμε τις εργασίες μας τώρα για την ομοθεσία περί ιδιωτικότητας και πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά και να βρούμε λύσεις οι οποίες θα είναι οι καλύτερε δυνατέ. Θα πρέπει βεβαίω να είμαστε σε επαφή, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ε, κάτι θετικό προς όλες τις κατευθύνσεις και για τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και για την ασφάλεια και για τον κανονισμό για την ε, ε, ιδιωτική, προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ευχαριστώ. Η Άννα Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργή που είστε εδώ. Εσείς επικεντρωθήκετε στην ασφάλεια των συνόρων, αλλά οι τρομοκρατικές επιθέσεις που βιώνουμε Ε, διαπράττονται από τους δικούς μας τους τρομοκράτες, εγχώρια προϊόντα. Επομένως ε, γίνεται εντό συνόρων. Γιατί λοιπόν δεν προσέχουν οι κυβερνήσεις ε, τα θέματα αυτά και δεν επικεντρώνονται σε μέτρα για να προλάβουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και να σταματήσει να προωθεί τη ριζοσπαστικοποίηση στα σοφρονιστικά καταστήματα που είναι σχολές ριζοσπαστικοποίησης γιατί να εισάγουμε ημάμιδες από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν και γιατί να μην ε, ευνοούμε ε, ημάμιδες που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ και έχουν εκπαιδευτεί εδώ που ε, δεν θα κάνουν και τέτοιας μορφής προσιλητισμό. Επίσης, γιατί παραβλέπετε όλοι δηλαδή εσείς οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων τις ε, εγκληματικότητα που έρχονται από αυτές τις χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων ε, μέσω της οποίας προσφέρεται εθνικότητα στους ανθρώπους που ξεπλένουν χρήματα. Γιατί δεν είναι η οδηγία για την ε, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων στην κορυφή των προτεραιοτήτων τα διότι και αυτό βοηθά για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή της και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό. Και επίση, γιατί δεν προωθούμε ασφαλεί και νόμιμε οδού για του μετανάστε και του πρόσφυγε, ώστε να μπορούν να κάνουν αίτηση να έρθουν εδώ και να μην τροφοδοτούμε το οργανωμένο έγκλημα και τους διακινητές ε, που είναι αυτοί οι οποίοι στην ουσία διαχειρίζονται τις ροές. Ευχαριστώ η Παρμπάρα Σπινέλη. Ευχαριστώ τους δύο υπουργούς για την παρουσία τους εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ε, αμφιβολίες ε, υπό το φως και των πρόσφατων επιθώσεων και την εθνικότητα των δραστών. Η πρώτη αμφιβολία, η διάθεση να ενισχύσουμε την προστασία των συνόρων συγχαίουμε εδώ την τρομοκρατία με το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων. Ζητάμε ενίσχυση του Frontex, ζητάμε να γίνονται ασκήσεις προσωμείωσης ε, για να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στη μαζική άφηξη μεταναστών. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι απάντηση στην τρομοκρατία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη μορφή τουλάχιστον της τρομοκρατίας. Δεύτερον, το ΕΤΙΑΣ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών, ε, το οποίο είναι στα σκαριά αυτή τη στιγμή ε, για να ελέγχουμε κάποιους πριν έρθουν στο χώρο Σέγγεν. Θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει την επαλήθευση πρώτης άφηξης και πώς. Η άλλη αμφιβολία που έχω είναι ο έλεγχος του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών. Αναφέρεστε στην ανάγκη να τηρήσουμε κάποιες υποχρεώσεις, λέγεται ότι το σύστημα Telegram δεν είναι αντίστοιχο με το WhatsApp, αλλά μόλις ε, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το ε, Telegram θα, αρχίσει να, θα γεννηθεί ένα άλλο που δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Επομένως το να ε, δέχεται κανείς τον έλεγχο δεν νομίζω ότι είναι η πλέον κατάλληλη λύση. Και κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω, και δύο αυτή τη στιγμή είστε στη διαδικασία προεκλογική εκστρατεία στη χώρα σα. Θα ήθελα να ρωτήσω το Γάλλο Υπουργό, για παράδειγμα, εάν όλα αυτά τα μέτρα ελέγχου των συνόρων δεν είναι λίγο μια αντιγραφή των θέσεων της ακροδεξιάς ε, στη Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Κοντεύουμε. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω καταρχάς για το θέμα της βιομηχανίας αυτής της παράνομης μετανάστευσης, της ε, λαθρέας μετακίνησης ανθρώπων, γιατί είναι πραγματικά ανησυχητικά τα στοιχεία τα οποία ακούμε από την στα. Ε, Θα θέλαμε λοιπόν και της πόλου. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι υπουργοί Προσφάτως λάβαμε πολλές πληροφορίες από το Ισραήλ και το Ισραήλ το γνωρίζει αυτό το, θέμα κατεξοχήν. Έχουμε πληροφορίες λοιπόν από υψηλόβαθμες ε, μυστικές υπηρεσίες και από αξιωματούχους ε, των μυστικών υπηρεσιών και συνταξιβετημένους και εν ενεργεία, οι οποίοι και μας ε, ενημερώνουν ότι η οδοί αυτή ε, μετανάστευσης χρησιμοποιούνται για να διοικητεύσουν τρομοκράτες στην Ευρώπη μας. Προειδοποιούν λοιπόν και μας ενιστούν να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή και να ελέγχουμε καλύτερα τις οδούς αυτούς, αυτές. Κάτι άλλο που αφορά και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα περιμένετε από τους συναδέλφους σας, τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, σε ό,τι αφορά την ε, ευθύνη, την νομική ευθύνη των όσων προσχωρούν στην ε, ISIS. Γιατί θα πρέπει να έχουμε και άλλα νομικά μέσα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται μόνο λες και συμμετέχουν σε στρατό άλλης ε, χώρας. Πρόκειται για προδοσία. Είναι εντελώς διαφορετική κατηγορία εγκλήματος και χωρίς προληπτικά μέτρα δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τέτοιες δραστηριότητες, ούτε να πείσουμε τις οικογένειές τους να τους ε, αποτρέψουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεφέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριο Σφερό. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα Ε, μάλιστα κυκλοφορεί τώρα και ένα βιβλίο Bienvenue Plus ε, ε, μπουβό όπου δύο ε, δημοσιογράφοι δυστυχώς δεν ακούγεται ο κύριος Φεραόν δυστυχώς οι διερμηνείς έχουν πρόβλημα δεν ακούμε τον κύριο Φεραόν δεν έχει ανοιχτό μικρόφωνο Να ξαναρχίσω λέει ο κύριος Φεραόν Έλεγα λοιπόν κύριε Υπουργέ ε, είπατε ότι διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ε, ιδιωτική ζωή, αλλά ε, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή γίνεται ένα σεισμός αποκαλύψεων. Υπάρχει το βιβλίο Bienvenue plus Bimont, όπου αριστεροί δημοσιογράφοι καταγγέλουν ένα σύστημα παρακολούθησης των υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές. Επομένως, ο διαχωρισμός εξουσίας ε, η καταπολέμηση των ε, καταχρήσεων και όλα αυτά είναι πολύ ωραία λόγια, αλλά ε, έχουν δείξει πολύ με το δάχτυλο τις υπηρεσίες των οποίων σήμερα είστε επικεφαλής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό. Και σε αυτήν την περίπτωση της γαλλικής, των γαλλικών εκλογών, των προεδρικών εκλογών, μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξουν ε, τέτοιου ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Μωράες, για, την, για τον χρόνο σας. Κρατήσατε, είστε πάρα πολύ αυστηροί με τον χρόνο και επομένως έχουμε την δυνατότητα τώρα να δώσουμε το λόγο στους υπουργού, Θα δώσω το λόγο πρώτο στον κύριο Τομάς Ντεμεζιέρ, παρακαλώ. Αγαπητέ Κλοντά, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι τόσο απλό τόσο γρήγορα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Να προσπαθήσω παρόλα αυτά. Ζητώ κατανόηση. Ενδεχομένω να μην ε, καταφέρω να δώσω όλε τι αποχρώσει. Καταρχά για την κυρία Μετσόλα. Για τη ΣΥΠΑ. Οι ΗΠΑ παίζουν ρόλο κλειδί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και κυρίως ε, οι νικητρίες δυνάμεις ε, των ΗΠΑ δεν έχουν επιτευχθεί από κανένα, καμία ευρωπαϊκή χώρα. Και είναι και αμφιλεγόμενα βέβαια, οι αμφιλεγόμενες οι μέθοδοι. Αλλά λόγω δεν είναι σαφές τι γίνεται με τις υποδείξεις των ΙΠΑ και σε ό,τι αφορά την αποτροπή επιθέσεων στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι προς το συμφέρον μας η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, προς το συμφέρον της Ευρώπης. Και εδώ υπάρχουν δύσκολα ζητήματα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή των δεδομένων. Αλλά να σας πω ότι με τη νέα α, κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ, τουλάχιστον για τη Γερμανία δεν ξέρω τι λέει ο Ματίας, δεν υπάρχει περιορισμός σε καμία περίπτωση της επικοδομητικής στάση στη συνεργασία, παρά το γεγονό ότι κάποιε στιγμέ ε, υπάρχουν επικρίσει κατά τη Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία, κανένα περιορισμό όμω τη συνεργασία και του επικοδομητικού πνεύματο σε ό,τι αφορά τι διάφορε ταυτότητε. Και στη Γερμανία, ξέρετε. Μέχρι το 2015 ούτε τεχνικός πόσο, ούτε νομικός πόσο όμως ήμασταν σε θέση να εξακριβώσουμε αν κάποιος, για παράδειγμα, ε, εμφανιζόταν στην κολονία, να διαπιστώσουμε ότι στη συνέχεια ε, βρισκόταν, για παράδειγμα, στη Στουρκάρδη. Δεν ήταν τεχνικός και νομικός ε, δυνατόν. Αυτό όμως άλλαξε και έτσι λοιπόν εντοπίζονται τις διαφορετικές ταυτότητες για τα βιομετρικά στοιχεία. Εδώ έχουμε να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα, αλλά να επισημάνω κάτι που είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο και σίγουρα θα σα ενδιαφέρει. Το θέμα των δακτυλικών αποτιμωμάτων και των βιομετρικών στοιχείων των ανηλίκων. Υπάρχει μια ηλικία κατά την οποία δεν έχει νόημα να συλλέγονται τέτοια στοιχεία γιατί βιολογικός πώ δεν ε, στέκουν. Αλλά πολλοί ανήλικοι δεν είναι καν ανήλικοι ουσιαστικά. και εκ παραλίλου υπάρχουν ε, και όρια σε ό,τι αφορά το τι είναι λογικό και τι είναι αναλογικό. Μπορούμε βέβαια, εντάξει, να καταγράφουμε και τα κόκαρα, τα οστά του ανθρώπου, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα και έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα των ανηλίκων και τη διαπίστωση της ηλικία ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις εθνικές ε, ευαισθησίες. Η κυρία Ζίπελ, συμφωνώ μαζί σας. χρειαζόμαστε για να είναι διαλειτουργικά τα συστήματα, χρειαζόμαστε και ενιαίους ορισμούς, όχι μόνο για το ότι είναι επικίνδυνο. Αλλά και για άλλα στοιχεία. Και αυτά θα πρέπει να αλλάξουν στο ΣΥΣ. Και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις διάφορες αρμοδιότητες στα κρατημέλη για να δούμε ποια υπηρεσία έχει πρόσβαση που. Αυτό, αν θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να υπάρχει κοινή δυνατότητα και περιορισμός πρόσβαση και μάλιστα δεσμευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι το τίμημα του, της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης για το ΣΥΣΕ που δεν αξιοποιήθηκε γέρος. Έχετε ένα δίκιο. Δεν είχε όμως καταγραφεί, δεν έχουν καταγραφεί τα στοιχεία επαρκώς. Δεν ήταν καλή λοιπόν η διαμόρφωση και πολλές αλλαγές κάναμε. Θέλαμε να βελτιωθεί το σύστημα λοιπόν και βελτιώθηκε πολύ, αλλά δεν είναι ακόμα επαρκής η βελτίωση. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών νομοθεσιών, αν προσέξουμε και τα ζητήματα διαλειτουργικότητας, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τέτοιων μέσων για τα δεδομένα αυτά. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, όχι της ε, Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αλλά θεωρώ ότι πολλά δεν έχουν νόημα για την κρυπτογράφηση. Να πω δύο λόγια για τους Βέλγους συναδέλφους. Να τους πω ότι εμείς στη Γερμανία δεν έχουμε προσωπικά εισιτήρια στο τρένο, με όνομα δηλαδή, και στο λεωφορείο και άρα τεχνικώς πώς δεν θα ήμασταν σε θέση να έχουμε κάτι αντίστοιχο με το PNR και να κάνουμε αντίστοιχους ελέγχους. Κάθε μέρα έχουμε 4 έως 5 εκατομμύρια άτομα τα οποία παίρνουν το τρένο στη Γερμανία χωρίς να υπολογίσουμε καν τα λεωφορεία. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς θα ήταν αναλογικό ένα τέτοιο μέτρο για την ερώτηση τη κυρία Ιντφέλτ για το τι συνέβη τελικά στο PNR. Δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία μέχρι το 2018 και δεν ξέρω ποια χώρα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Εμεί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέχρι το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται και η θητεία τη γερμανική κυβέρνηση. Ήταν πολύ ωριακό, ωριακή η προθεσμία και η Γερμανία θα τηρήσει, ελπίζω και όλοι οι υπόλοιποι, την προθεσμία. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πιο πολλές πληροφορίες. Να πω δύο λόγια για το... για το θέμα του άμρι. Αν ξέραμε ότι ο άνθρωπος αυτός ε, είχε καταθέσει αυτή την αίτηση ασύλου στην Ιταλία και ότι είχε πάει στην Ιταλική ε, φυλακή, αυτό δεν είναι θέμα ότι δεν το ξέραμε, ότι δεν το χρησιμοποίησαμε ως στοιχείο, δεν το ξέραμε. Αυτό λοιπόν είναι θέμα το ότι θα πρέπει να κάνουμε εμείς οι υπουργοί. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν ποινικοί. Ε, οι ποινικές διαδικασίες για τη βελτίωση των ε, διαδικασιών αυτών. Κάτι που είπαν και οι Γάλλοι συνάδελφοι. Και η κυρία Γκόμες γιατί αναφέρετε τόσο περιορισμένα το σκέλος της πρόληψης. Πολύ δικαιολογημένη ερώτηση, αλλά να σας πω το εξή. Μια μικρή παρατηρήση. Καταρχάς, σε πολλά κράτη δεν είναι υπουργοί α, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το σκέλος της πρόληψης. Αυτό φυσικά δεν είναι δικαιολογία, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι τα τελευταία χρόνια συζητείται πάρα πολύ το θέμα τη πρόληψη. Παλιά ξέρετε το θέμα του Υπουργού Εξωτερικών και της ε, δικαιοσύνη και ε, των ε, αστυνομ... της αστυνομίας ήταν ε, πάρα αργά. Δεν θεωρούνταν τόσο σημαντικά. Αυτό έχει αλλάξει. Και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία ήταν πάρα πολύ δυναμική στην καταπολέμηση τη Δημοκρατία, ήταν η χώρα η οποία ήταν πιο δυναμική στο σκέλο τη πρόληψη. Και αυτό έχει να κάνει και με το διαδίκτυο η Γαλλία και η Γερμανία ανέλαβαν μια πρωτοβουλία η οποία παρουσιάστηκε και στο Συμβούλιο για τα πολλά δίκτυα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Από όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να συνθέσουμε ένα ευρωπαϊκό κέντρο για την πρόληψη, για να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη στις εργασίες αυτές, να υπάρχει σωστός συντονισμός και βελτίωση. Το είπα και στο Συμβούλιο ότι δεν είναι δυνατόν να έχει αυτή τη στιγμή καλύτερη δικτύωση, ε, μία σπήρα δολοφόνων από ότι τα εθνικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κυρία Έρνστ τώρα. Τη γνωρίζουμε τη συζήτηση αυτή και από το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Τα μέτρα αυτά δεν ε, οδήγησαν σε πρόληψη της επίθεσης, άρα δεν έχουν νόημα. Κοιτάξτε, έγιναν επιθέσεις στη Γαλλία, όπου οι δράστες δεν κατέφθασαν με αεροπλάνο. Αλλά υπήρχαν επιθέσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν τα αεροπλάνα. Και τέτοια μέτρα δεν έχουν να κάνουν συχνά μόνο με την πρόληψη των ενεργειών αυτών, αλλά και για την διευκρίνηση και την επίλυση και την, τον, τον εντοπισμό δικτύων α, για τις διακραγωγή των επιθέσεων. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν σημείο. Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη δικτύωση μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Και οι μυστικές υπηρεσίες, θα ήθελα να προσθέσω, θα μπορούσαν να δικτυωθούν καλύτερα. Αλλά αυτό φαντάζομαι δεν σας βρίσκει σύμφωνος όλους σε ό,τι αφορά τη δικτύωση των μυστικών υπηρεσιών. Εγώ είμαι μάλλον διστακτικό σε ό,τι αφορά κάποια κράτη, αλλά η δικτύωση των αστυνομικών υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο είναι εκ των ΟΚ άνευ και η κοινή έρευνα. Και να σας πω ότι η εκτίωση της αστυνομία δεν ε, αντικαθιστά την ε, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Είπατε ότι η αρχή ο ορισμός της δημοκρατίας ε, θα πρέπει να είναι κοινό. Το ποινικό δικαίωμα είναι φυσικά εθνική αρμοδιότητα, αλλά με τον ΟΙΑ αποφασίσαμε και δημιουργήσαμε πολύ, καλούς, πολύ καλές νομικές βάσεις για τον ορισμό της τρομοκρατίας, για την τρομοκρατική οργάνωση. Η τρομοκρατία ως όρος δεν νομίζω ότι είναι ε, δύσκολο να οριστεί, αλλά η επικινδυνότητα θεωρώ ότι είναι πιο ε, ουσιώδες ζήτημα για το τι θα μπει και πού, σε ποια βάση δεδομένων. Να πω ότι και η Γερμανία ήταν διστακτική σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τη, για δύο λόγους μάλιστα. Καταρχάς, γιατί είχαμε ήδη πολλούς ε, πρόσφυγες και κατά δεύτερον θέλαμε να υπάρχει relocation μόνο εφόσον ήμασταν βέβαιοι ότι όλοι αυτοί που ήταν στην Ελλάδα και στην Ιταλία είχαν καταχωριστεί. Ζητώ κατανόηση. Και φυσικά το θέμα της εφαρμογής του Δουβλίνου και στην Ελλάδα και εν μέρει και στην Ιταλία ως ε, Κρατήτη αποφασίσαμε να αλλάξουμε την τοποθέτησή μας και από τον Οκτώβριο, το φθινόπωρο, ε, δεσμευτήκαμε έναντι της ε, Ιταλίας και της Ελλάδας ότι κάθε μήνα θα κάναμε relocation για 500 άτομα. Και η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν αρκετά ικανοποιημένε. Η κυρία Χόλμαϊρ ζήτησε να διευκρινίσουμε κατά πόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα καταχώρηση των δεδομένων. Ναι, υπάρχει πρόβλημα καταχώρηση των δεδομένων στι βάσει και ιδιαίτερα κάποια κράτη διαμαρτύρονται ότι υπάρχει περιορισμένη εισαγωγή των δεδομένων. Ιδιαίτερα μια μεγάλη χώρα, την οποία ξεχνώ, αλλά έχει τον ε, διοικητή της Europol. Και θέσατε και ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα. Γιατί τέτοια δεδομένα είναι προληπτικά, χωρίς να πούμε ότι όλοι είναι υπογενική υποψία για το Eurodac για παράδειγμα. Εδώ πέρα να κάνω μία σύγκριση με το σύστημα πληροφόρηση για τις θεωρήσεις. Θέλουμε κάποιοι άνθρωποι να ταξιδεύουν χωρίς υποχρέωση θεώρησης και κάποιοι άλλοι υποχρεούνται να ζητήσουν βίζα. Κάθε αίτημα για χορήγηση θεώρησης ελέγχεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας για το κατά πόσο υπάρχει κάποια υποψία δεν είναι μια γενική γενικευμένη υποψία, είναι θέμα μέτρου πρόληψη. Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη Γυροντάκα. Με την κυρία Ρεβό. Έθεσε μια πολύ μια ερώτηση Άμα, για το κατά πόσον το ζητάμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από το Συμβούλιο. Γιατί προσπαθούμε να μην ε, πιέζουμε τους συναδέλφους, αλλά να τα ρίχνουμε αυτό στην Επιτροπή. Η επιστολή αυτή τι έλεγε. Όχι να εφευρεθούν νέα στοιχεία, αλλά να εφαρμοστούν γρήγορα τα όσο ήδη είχαμε αποφασίσει για την εκπαίδευση τώρα των υπαλλήλων. Σίγουρα μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά ελπίζω κάθε αστυνομικό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να έχει την κατάρτιση να ελέγξει ένα διαβατήριο, να ελέγξει ένα αρχείο και σε ό,τι αφορά τη Frontex φυσικά έχουν ειδική εκπαίδευση. Εναρμόνιση ναι, αλλά αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να υπάρχει επαρκές προσωπικό για τη Frontex, γιατί αν περιμέναμε να υπάρχει σωστή και κοινή εκπαίδευση, αυτό θα αποτελούσε δικαιολογία για πολλές χώρες, ε, ότι δεν έχουμε ακόμα κοινό σύστημα εκπαίδευση και δεν θέλαμε να δώσουμε αυτή τη δικαιολογία σε κανέναν. Η κυρία Βίξτρομ σε ό,τι αφορά την τρομοκρατία, έθεσε το ζήτημα με τη μετανάστευση. Είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα αυτό, ξέρετε. Και θα πρέπει να γίνει διαχωρισμό εδώ. Οι πιο πολλοί πρόσφυγες είναι θύματα, δεν είναι θύτες. Φυσικά, είναι γεγονός ότι μεταξύ των προσφύγων έχουν περισφρήσει και τρομοκράτες. Σκόπιμα ενδεχομένω ε, για να αφήσουν ίχνη, για παράδειγμα, στο Στάντεφ Χάνσε όπου έγινε η επίθεση, θεωρούμε ότι ήταν ε, τεχνητά τοποθετημένη αυτή η ένταξη για να προκαλέσει ακριβώς τη συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ του διαχωρισμού της ε, μετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Όπου υπάρχουν φυσικά ε, σύνδεσμοι και σημεία επαφής θα πρέπει να τα αναφέρουμε και να τα συζητούμε. Το βασικό θέμα το οποίο δεν θα επιλύσουμε σήμερα έχει ουσιαστικά καταληφθεί το Δουβλίνο. Τι θα κάνουμε στο μέλλον λοιπόν για το θέμα αυτό. Και αυτό αποτελεί τμήμα του συμβιβασμού μεταξύ Γαλλία και Γερμανία για το κοινό σύστημα ασύλου. Προτείνω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε και να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ μικρών, μεσαίων και μεγάλων α, όγκων. Υπήρχε μια οδηγία η οποία, ε, για μαζική εισρωή, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε παρά το γεγονό ότι υπήρξε μαζική εισρωή. Άρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει άλλη νομοθεσία για το κατά πόσον μιλάμε για μικρό, μεγάλο ή μεσαίο όγκο εισρωής ε, μεταναστών. Τέθηκε και το ερώτημα για τα βιομετρικά δεδομένα και κατά πόσον μπορούν να βελτιωθούν στις εθνικές ταυτότητες. Καλή ερώτηση. και το κοιτάμε σε ό,τι αφορά την ελευθερία από το καθεστώ των θεωρήσεων. Λέμε σε κάποιε χώρε ότι μπορείτε να, είσαστε, να πάρετε απαλλαγή μόνο αν έχετε βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήριά σα. Πολιτική πίεση μένα, αλλά εν πάση Το κάνουμε. Είναι σωστό μέτρο, θεωρώ. Και ίσω ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εδώ. Ύστερα, θέλετε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα αν έχουμε μια δυναμική, ένα δυναμικό IP address. Πώς μπορούμε εκ των υστέρων να κάνουμε και να αξιοποιήσουμε τα ονόματα. Θεωρώ ότι είναι θέμα κλειδί αυτό. Και αυτό που θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει είναι το εξή, αυτό που χρειαζόμαστε δηλαδή. Το συζητάμε και στη Γερμανία και θα πρέπει να το συζητήσουμε σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε, πιστεύω, ε, πληροφορία προέλευσης και για τις μυστικές υπηρεσίες και για ενημερώνουμε τους παρόχους ποιος χρησιμοποίησε τη διεύθυνση IP. Και σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο. Το θέμα της διαλειτουργικότητας. Ο κύριος Μπόνι ρώτησε τι γίνεται με την τεχνική διαμόρφωση. Έχετε δίκιο. Αυτό που δεν επιθυμούμε είναι να καταστούν όλες οι επενδύσεις στον τομέα του IT α, ε, ανούσιες. Δεν είμαι ειδικό για θέματα IT, αλλά θα ήθελα να πω ότι η έξυπνη οργάνωση των διεπαφών θα διευκολύνει την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Προ την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δουλέψουμε. Αυτό κάνει άλλωστε και η ομάδα υψηλού επίπεδου. Θέλουμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό. Η κυρία Γκόμε, πέρα από το θέμα τη πρόληψη, έθεσε και το ερώτημα του γιατί δεν ε, θέτουμε προτεραιότητα και το ξέπλυμα χρήματος. Κοιτάξτε, το κάνουμε, αλλά βασικά είναι αρμοδιότητα των Υπουργών Οικονομικών. Το κάνουμε πολύ στυλ. Και τέθηκε και το θέμα των παράνομων και νόμιμων οδών προς την Ευρώπη. Μεγάλο ζήτημα αυτό και δεν θα μπορέσουμε να το λύσουμε σήμερα. Το πρόβλημα είναι, ξέρετε ποιε είναι οι προτάσει που έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι. Και αυτό είναι, εδώ έγκυται και η διαφωνία, αν θέλετε. Νομίζω ότι αν δημιουργήσουμε νόμιμε οδού και δεν κλείσουμε τις παράνομες οδούς που χρησιμοποιούνται ως τώρα, θα πούνε πάνω-πάνω οι νόμιμοι μετανάστες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι νόμιμες οδοί για όσους χρήζουν βοήθειας και για τους οικονομικούς μετανάστες. Αντί για παράνομη μετανάστευση. Αυτό φυσικά είναι πιο εύκολο να το πούμε παρά να το υλοποιήσουμε, όπως το ξέρετε όλοι σας. Είπα δύο λόγια για το ποιος ελέγχει τώρα το αίτιας ή συνοριακές ε, αρχές ή αρχές που κάνουν τον έλεγχο και τις θεωρήσεις. Νομίζω ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν το αίτιας. Είπατε τώρα ότι για ένα τηλεγράφημα τον έλεγχο τον κάνει άλλη εταιρεία. Κοιτάξτε, αυτό δεν με πείθει επιχείρημα. Όλοι μαζί από κοινού για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια για την καταπολέμηση τη παιδική πορνογραφία. Στην αρχή ήταν. Ε, φαίνονταν χωρί τέλο αυτό ο αγώνα ε, και μάταιο. εν τω μεταξύ, έχει αλλάξει η κατάσταση. Έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Ούτε μπορούμε να λέμε ότι δεν έχει νόημα να καταπολεμούμε την παιδική φωτογραφία και τη μία συγκεκριμένη φωτογραφία γιατί μπορεί να εμφανιστεί κάποια άλλη κάπου αλλού. κύριος Γιούρεκ ζήτησε να το πούμε τι προσδοκίες έχουμε από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Έχουν γίνει λάθη. Αλλά αυτό που είναι σαφές και δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Αν κάποιος ε, είναι ο του Ισλάμ, δεν υπάρχει λόγος να δραστηριοποιηθεί ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Αν είναι Ισλαμιστή, τα πράγματα ενδεχομένω να έχουν διαφορετικά, διαφορετική βαρύτητα. Αλλά ούτε κάθε Ισλαμιστή ε, είναι τρομοκράτη. Πάλι υπάρχει διάκριση λοιπόν που πρέπει να γίνει μεταξύ των Ισλαμιστών, Ισλαμιστών τρομοκρατών. Σε ό,τι αφορά του υπουργού ε, δικαιοσύνη, είναι πιο πολύ το θέμα. Και να σα πω ότι σε ό,τι αφορά τι ποινικέ ε, διαδικασίε και τι ποινικέ διώξει, δεν είναι τόσο πολύ η ανταλλαγή δεδομένων στι στις άλλες περιπτώσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά τι απαντήσει μου. Αν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μη μιας ε, ε, ε, ε Αυτό σημαίνει ότι ίσως εσείς, κύριε Φέκλη, μπορείτε να είσαστε λίγο πιο σύντομοι. Σύντομος. Ό, κοιτάξτε, συμφωνούμε με πάρα πολλά πράγματα. Απίνθησε ο κοιτάξτε, συμφωνούμε με πάρα πολλά πράγματα. Ε, απήντησε ο συνάδελφός μου, ο κ. Ντεμεζιέρ, για τα πάντα, οπότε με έχει καλύψει σε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα απαντήσω σε κάθε μία ε, ερώτηση ξεχωριστά, αλλά ίσως θα δώσω κάποια επιπλέον στοιχεία. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση με τις ΗΠΑ, βεβαίως είναι μείζον ζήτημα το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών είναι αυτό που είναι ε, και όμως επί πολλών θεμάτων εξακολουθούμε να έχουμε εταιρικέ σχέσεις πολύ σημαντικές. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο πιο παλιός σύμμαχος της ε, Γαλλίας ιστορικά μιλώντας και βεβαίως και όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας και αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ μας ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ δεν έχω έρθει ακόμα σε επαφή με τον Αμερικανό ομολογό μου από την προηγούμενη Τετάρτη που ανέλαβα αλλά ε, οπωσδήποτε ε, συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα υπάρχουν, είναι σημαντικές, ε, είναι δυνατές και ε, σημασίας και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για το μέλλον οπωσδήποτε θα έχουμε ε, την δυνατότητα να εργαστούμε ε, σε αγαστή συνεργασία. Όσον αφορά την διαλειτουργικότητα και τις, ε, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Συμφωνώ απολύτως, συμμερίζομαι απολύτως αυτά που είπε ο Τωμάντε Μεζιέρ σχετικά με την απέτηση διαλειτουργικότητας. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, είναι ρεαλιστικό να δίνουμε στις ε, ομάδες επιβολής ε, του νόμου ε, δυνατότητες. Αλλά βεβαίως οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και βεβαίως δεν θα έχουν σαν αυτό σκοπό πάντα τον όλο και μεγαλύτερο έλεγχο. Όχι, θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη αξία και θα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να υπεραμεινθούμε των ιδεωδών και των αξιών μας. Επομένως, ό,τι χρειάζεται για την καταγραφή, για την ε, ε, διαβούλευση και για την, ε, για την χρήση και για την διατήρηση θα ισχύσουν. Και θα αντλούμε πληροφορίες κάθε φορά που αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης έγινε λόγος για το PNR των ταξιδιωτών ε, των σιδηροδρόμων. Εμείς ε, ε, δεν το βλέπουμε με άσχημο μάτι. Ας δούμε τι συνέβη στο τρένο Θαλής ε, που πήγαινε από το Άμστερνταμ στο Παρίσι. Δώσαμε λοιπόν επί της αρχής την σύμφωνη γνώμη μας για να ξεκινήσει ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα και γνωρίζετε ότι έχει δημιουργηθεί μια ε, task force, μια ομάδα εργασίας η οποία ε, θα ασχοληθεί με τη μελέτη αυτού του θέματος. Επίσης, ε, έγινε λόγος για την επίγουσα κατάσταση, δηλαδή, καθεστώς επίγουσας κατάστασης που ισχύει στη Γαλλία. Ε, εγκαθιδρύθηκε μετά από τις ε, πρώτες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και πρόκειται για μια διαδικασία, για ένα καθεστώς το οποίο προβλέπεται στο Γαλλικό Σύνταγμα. Επομένως, το Σύνταγμά μας προβλέπει την χρήση αυτού του καθεστώτος και μάλιστα αναφέρει και το πλησιώνει το καθεστώς αυτό με συγκεκριμένο τρόπο. Πρόκειται για μία από τις ε, συνταγματικές ε, αρχές ε, και το Συνταγματικό Συμβούλιο έχει δυνατότητα να κρίνει την νομιμότητα των πράξεων και να ελέγχει λοιπόν το καθεστώς. Αυτό το καθεστώς βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει ένα έκτακτο καθεστώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλες οι αρμόδιες αρχές κάθε φορά που κατέστη απαραίτητη η παράταση μέσα από ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο ε, οι αρμόδιες αρχές το έχουν ε, ε, ξαναπεί και το έχουν υπογραμμίσει. Παρατάθηκε για μία ακόμα φορά εν των προεδρικών εκλογών και λόγω της αύξησης της απειλής αυτή την περίοδο στη χώρα μετά από ψηφοφορία του Κοινοβουλίου. Και στους επόμενους μήνες οι βουλευτές θα αποφασίσουν εάν και κατά πόσον θα πρέπει να παραπτωθεί ακόμα μία φορά το καθεστώς αυτό. Πρόκειται πάντως για ένα καθεστώς το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα. Όσον αφορά τη Eurodax, συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο Τομάς Δεμεζιέρ. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ε, ε, θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε και το πνεύμα ε, το οποίο υπαγόρευσε την επιστολή μας προς το, την Κομισιόν γιατί πραγματικά θέλαμε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και πιστεύουμε ότι η υλοποίηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτική. Πολλές αρχές έχουν τεθεί, σημαντικές, ισχυρές αρχές ε, και ε, πιστεύουμε ε, ότι τώρα επί πολλών θεμάτων να περάσουμε, πρέπει να περάσουμε στην λειτουργική φάση έτσι ώστε να μπορέσουν και οι αρχές μας να δουλέψουν αποτελεσματικά. Μπορώ να συμφωνήσω για μία ακόμα φορά με αυτά που πολύ ορθά αναφέρθηκαν προηγουμένως όσον αφορά το Δουβλίνο και την ε, ε, relocation. Υπάρχει η συμφωνία, αναφέρθηκε αυτό. Απλώς να πω ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι οι δύο χώρες οι οποίες ε, έχουν, περισσότερο, έχουν κάνει τις περισσότερες επανεγκαταστάσεις, έχουν δηλαδή τους μεγαλύτερους αριθμούς από επανεγκατασταθέντες. Όλες οι χώρες φυσικά θα πρέπει να αναλάβουν τις, ε, ε να αναλάβουν ε, τις υποχρεώσεις τους. Όσον αφορά τώρα πλαστογραφημένα έγγραφα, ε, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει ακόμα ευρωπαϊκό πρότυπο, οπωσδήποτε αυτό θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Σε εθνικό επίπεδο στη Γαλλία εμείς έχουμε βιομετρική βάση για, τα, για τις ταυτότητες, η οποία λειτουργεί καλά, είναι επιχειρησιακά άρτια όσον αφορά το θέμα των ξένων ημάμιδων. Είχαμε μια πολύ θετική συζήτηση πριν από λίγο ε, στο Συμβούλιο ε, Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ε, όσον αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και εμείς ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες μέλη να κινητοποιηθούν ακόμα περισσότερο ε, και επομένως συμφωνούμε απολύτως ότι πρέπει ε, το Συμβούλιο κατά της ριζοσπαστικοποίησης να γίνει ευρωπαϊκό μέσο, ευρωπαϊκό εργαλείο και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς ε, για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και επομένως και την καταπολέμηση αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Να σας πω επίσης ότι στη Γαλλία κυρίως λόγω του καθεστώτος ε, επίγουσας κατάστασης έχουμε κλείσει σαλαφιστικές, ε, σαλαφιστικά τζαμιά ε, όταν υπήρχαν οι προϋποθέσεις οι νομικές για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο προκάτοχός μου, ο, ο κύριος Λερού, αλλά και πριν από αυτόν ο κύριος Κασνεύ, είχαν δουλέψει με πολύ αποτελεσματικό και απαιτητικό τρόπο πάνω από 20 τέτοια τζαμιά έκλεισαν ε, και συνεχίζουμε ε, με πλήρη επαγρύπνηση ανα πάσα στιγμή παρακολουθούμε ε, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια το τι, το τι συμβαίνει στο γαλλικό έδαφος. Οτιδήποτε συμβαίνει στη γαλλική επικράτεια θα πρέπει να σέβεται τους γαλλικούς νόμους. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά αυτές τις μαύρες ε, προπαγάνδες, ε, ε, όλοι πολύ εύκολα έχουμε την καραμέλα του πατριωτισμού ε, ε, στο, στόμα, αλλά η πραγματικότητα τελικά είναι διαφορετική. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπήρξε πάρα πολύ σαφής σήμερα και μπορώ να σας πω ότι και από πλευράς του Υπουργείου των Εσωτερικών δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς ενστερνιστήκατε στοιχεία τα οποία δεν έχουν ε, επιβεβαιωθεί και μάλιστα και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου ε, λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ε, που να επιβεβαιώνουν ότι όντως υπάρχει ένα μαύρο γραφείο, ένα μαύρο καμπινέ υπουργών Ευχαριστώ. Ξέρω κύριε Υπουργέ Ντεμεζέρ ότι πρέπει να φύγετε, μας το είπατε αυτό αλλά πάντα συζητιέται εδώ στην Επιτροπή. Ξέρω ότι έφυγαν και κάποιοι συνάδελφοι, αλλά θα αναγνωρίσουν ότι πάντα το συζητάμε και υπάρχει και μια ε, ένταση, αν θέλετε, για το κατά πόσον ε, θα καλούμε τους ε, ε, υπαργούς εσωτερικών εδώ να τα συζητάμε απευθείαν, εσύ απλώς θα συζητούμε απλώς με την Προεδρία. Νομίζω ότι η σημερινή ημέρα αποδεικνύει ότι αξίζει τον κόπο να γίνεται μια διεξοδική συζήτηση και μάλιστα όταν είναι καλά δομημένη μπορεί να γίνει κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων. Προφανέστατα υπάρχει και ε, διαφορετική ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και εσάς ε, και τη γραμματέα της Επιτροπής μας που τα οργάνωσε όλα αυτά και σας ευχαριστώ και που ήσασταν και τόσο πειθαρχημένοι όλοι με το χρόνο. Κυρία Σίπελ, θέλετε να κάνετε και δεύτερη ερώτηση. Πολύ σύντομα, διότι ο κύριος Ντεμεζιέρ στην αρχή είπε ότι θα επανέλθει αργότερα στο θέμα της κρυπτογράφησης και της κωδικοποίησης, αλλά μου διέφυγε. Επαναλαμβάνω. Εγώ είμαι υπέρ της κωδικοποίησης ε, end-to-end, σε διαφορά τις ε, επικοινωνίες. Αυτό μάλιστα το παροτρύναμε, το ενθαρρύναμε. Γιατί θέλουμε οι μεταφορές αυτές να είναι ασφαλείς. Και σίγουρα θα χρειαστούμε ασφαλή επικοινωνία για την ψηφιοποίηση 4,0. Δεν θα έχει επιτυχία το σύστημα αν αρχίσουμε και ανησυχούμε για το κατά πόσο είναι ασφαλής η σύνδεση. Σε ό,τι αφορά για παραπαραγγελίες, σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες με τις ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Αλλά δεν είναι δυνατόν αν σήμερα υπάρχει δυνατότητα υποκλοπής μιας ε, τηλεφωνικής συνομιλίας ε, και όντως παρακολουθείτε μια μια... ένα τηλεφώνημα μέσω κινητού τηλεφωνίου, τηλεφώνου, να μην υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα ο πλευρά κράτου δικαίου αν η κλίση αυτή λαμβάνει η χώρα μέσω Skype. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώ σε τέτοιε περιπτώσει μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά. Το πρώτο πρόβλημα είναι κατά πόσον καταγράφεται μια συζήτηση WhatsApp ε, και μπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε αυτή αναδρομικά, όχι μόνο το τι έγινε η συνομιλία, αλλά και το τι περιλάμβανε η συνομιλία. Αλλά αυτό που είπατε επί της αρχής είναι ότι η υποκλοπή τηλεφωνημάτων, για παράδειγμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιτρέπεται, αλλά δεν είναι δυνατόν η αστυνομία, μη λαμβάνοντα υπόψη τα κριτήρια αυτά, να παρακολουθεί πέρα από το προσωπικό επίπεδο ασαφή αριθμό ατόμων. Συμφωνώ σε αυτό. Δεν υπάρχουν πιο πολλά τα δικαιώματα αλλά ούτε και πιο λίγα. Και από τεχνική απόψη το ξέρει και ο Γάλλο συνάδελφο ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τεχνικέ ε, λύσει και καλύτερα να γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά. Με το είπατε εσεί, αλλά το λένε και εγώ δεν συμφωνώ. Όταν ε, λένε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να ψάχνουμε στο Darknet για εμπορικό όπλων, για παιδική πορνογραφία. Αυτά δεν ισχύουν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επερωτηση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να βρεθώ στο δρόμο ενός ε, Γερμανού Υπουργού και το τι γίνεται με κρυπτογράφηση. Πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση για την ε, κρυπτογράφηση και το τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και που απαντήσατε στην επιπλέον ερώτηση. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφου για τις ερωτήσει τους και τους Υπουργού για τις πληροφορίες. Θα συζητήσουμε το Συμβούλιο Υπουργών ε, Δικαιοσύνης ε, και Εσωτερικών Υποθέσεων την Πέμπτη. Σα ευχαριστώ και σας που βρήκατε το χρόνο να έρθετε. Σα ευχαριστώ πολύ.